Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχουμε τον εισηγητή μαζί μας, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλοι σας είστε πολύ σημαντικοί, αλλά πάνω απ' όλα εισηγητής. Το πρώτο μας σημείο στην απόψινή μερίσια διάταξη είναι η μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρήπων και η τροποποιητική οδηγία 2003-35. Θα ήθελα να σας πω ότι η ΤΡΕ έκανε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 μετά από την παρουσίαση της Επιτροπής για τις δύο νομοθετικές προτάσεις όσον αφορά την ποιότητα του αέρα και τις βιομηχανικές εκπομπές. Στο πρόγραμμα εργασίας της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει ότι θα απέσυρε την πρόταση περί εθνικών εκπομπών, αλλά μετά από την επιμονή των κρατών μελών και του Ευρωκοινοβουλίου, το, η Κομισιόν αποφάσισε να το διατηρήσει στην ημερήσια της διάταξη το θέμα αυτό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι Μιλάμε για απλοποίηση, για επικουρικότητα, για τις δυνατότητες των κρατών μελών, αλλά τελικά θέλουμε να τα μελετούμε όλα και να αποφασίζουμε επί παντός επιθετού. Και αυτό είναι ένα πολύ σχετικό παράδειγμα. Σήμερα η εισηγητής θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του. Δεν είναι υπεύθυνο για ολόκληρο το σχέδιο, αλλά θα περιμένουμε την ε, δική σας νόμη, συνάδελφε Γερέκα, και οι υπόλοιποι θα έχετε τη δυνατότητα να παρουσιάσετε τις γνώμες σας, τις απόψεις για αυτό το σημαντικό θέμα. Ως ήρθιστε, θα ξεκινήσουμε με τον εισηγητή μας, τον κύριο Άνταμ Γκέρεκ. Κύριε Γκέρεκ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και θα ήθελα να σας πω ότι είμαι πολύ ευτυχής που το θέμα, ανεξάρτητα από το τι σχέδια έχει η Επιτροπή ή την έλλειψη σχεδίων, είμαι ικανοποιημένος που το θέμα παρέμεινε στην ατζέντα της Κομισιόν. Ποιος είναι ο στόχος της νέας οδηγίας. Σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο της 18 Δεκεμβρίου, για την μείωση των εθνικών εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρήπους, και την τροποποίηση της οδηγίας του 2003, ο στόχος είναι να παροτρινθεί η καινοτομία που μπορεί να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη αλλά και που θα οδηγήσει στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης καθώς και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Τα κράτη-μέλη έχουν συγκεκριμένα όρια εκπομπών. Η βασική τροποποίηση σε σχέση με την οδηγία του 2003 συνίσταται στην εισαγωγή του μεθανίου αλλά και στην εισαγωγή διαβουλεύσεων περί των επενδύσεων που στο μέλλον θα μπορούν να συνδέονται με τις εκπομπές. Το σχέδιο δεν περιλαμβάνει όλες τις εκπομπές, κυρίως στερεών σωματιδίων κάτω από τα 2,5 ε, μικρό, μικρό και δεν υπάρχουν δεν συμπεριλαμβάνονται μάλλον οι πολυχλωρινωμένοι υδρογονάνθρακες. Επίσης, δεν αναφέρεται το πολύ χαμηλό είχα πολύ χαμηλές εκπομπές που είναι πολύ ε, προβληματικές ιδιαίτερα για τους κατοίκους κάποιων νέων κρατών μελών που όπως η Πολωνία ε, κάποιες φορές η ε, ρήπη όπως το, το διοξίδιο του θείου ε, δεν αναφέρονται. Τέτοιου είδους ρήποι εκπέμπονται στην διάρκεια εξόριξης, για παράδειγμα. Ε, ή, επίσης, κατά τη μεταφορά πετρελαίου εκπέμπονται αυτό το, αυτός ο ρήπος. Με αυτήν την πρόταση εισάγονται διαφορές για τα διάφορα κράτη-μέλη όσον αφορά την αναφορά ε, για τους ρήπους, γιατί είναι δύσκολο να εφαρμοστούν τα ίδια κριτήρια για όλα τα κρατημέλη. Τα όρια εκπομπών για τα κρατημέλη μπορεί να αναφέρονται στις εκπομπές που είναι μετρήσιμες και μπορούν να ε, καταμετρηθούν, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εκπομπές που είναι δύσκολο να μετρηθούν αλλά ξέρουμε πως αυτό ισχύει για τα νανοσωματίδια στην ατμόσφαιρα γιατί ο αριθμός τους αυξάνεται και είναι επικίνδυνα διότι μπαίνουν στο σώμα μας και μπορεί να είναι καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Ίσως γι' αυτό να έχουμε αυξανόμενα περιστατικά καρκίνου των πνευμόνων. Δεν έχει αναλυθεί όμως, δεν έχουν αναλυθεί αυτά τα στοιχεία. Πάντως μπορούμε να περιορίσουμε τα όρια για τις εκπομπές και δε, επίσης δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η επιρροή τους στις κλιματικές αλλαγές γιατί ε, αυτά είναι συστατικά των διαφόρων αεροζόλ. Ε, η έννοια επίσης της χρήσης των ε, πτυτικών χημικών συστατικών ε, είναι κατά προσέγγιση διότι μπορεί να υπάρξει εκπομπή αυτών στην ατμόσφαιρα και οι δικοί της Κομισιόν θα έπρεπε να τα ορίζουν καλύτερα και να μας παρέχουν και τρόπους παρακολούθησης ή καταμέτρησης. Επίσης η αποσύνθεσή τους ε, είναι σημαντικό στοιχείο. Αυτά τα νοσοματίδια εκπέμπονται από τις, ε, τους κινητήρες δίζελ. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τα όρια γιατί ο αριθμός των αυτοκινήτων με κινητήρα δίζελ αυξάνεται στην Ευρώπη. Τα στοιχεία λοιπόν δεν είναι πια ενήμερα. Έχω επίσης και κάποια επίσης, τυπικά προβλήματα για το κείμενο, ιδιαίτερα όταν αυτό αναφέρεται σε διάφορα παραρτήματα που δεν είναι πλέον δεσμευτικά. Έχω την άποψη ότι αν το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θέλουμε να εγκριθεί ως οδηγία, θα πρέπει να φέρει τα δικά του παραρτήματα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρόνο σας. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Εξ ονόματος του ΕΛΚΑ, η κυρία Βίρκουνεν. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκέρεκ για την προπαρασκευαστική εργασία του. Νομίζω ότι ήταν ε, κάπως καλύτερη η αρχική ιδέα της Κομισιόν. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί αυτή η οδηγία για να εξετάσουμε μαζί πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε 32 ενεργειακούς στόχους και πώς μπορούμε να καταργήσουμε περί τη νομοθεσία. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν καλή ιδέα της Κομισιόν να αποσύρει αυτή την οδηγία και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους ενεργειακούς μας στόχους. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι σημαντική η μείωση των εκπομπών. Θετικό εδώ είναι ότι στόχος είναι η αποτελεσματικότητα και ότι τα κράτη-μέλη μπορούν μόνο τους να αποφασίσουν πώς θα μειώσουν τις εκπομπές και τι μέτρα θα χρησιμοποιήσουν για να το πετύχουν αυτό. Πρέπει όμως να φροντίσουμε η οδηγία να μην επιβάλλει επιπλέον άχθος ε, στην βιομηχανία. Ιδιαίτερα κάποιοι βιομηχανικοί τομείς ε, αντιμετωπίζουν σημαντικό άχθος. Βλέπουμε σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και θα πρέπει να φροντίσουμε αυτές να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσει. Ο στόχος για το 2025 δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι δεσμευτικός αυτή τη στιγμή. Εάν έχουμε ενδιάμεσους δεσμευτικούς στόχους, αυτό μπορεί να εμποδίσει την θετική αποδοχή του όλου πακέτου. Και φυσικά θα πρέπει να φροντίσουμε από το 2020 μέχρι το 2030 να έχουμε αποτελεσματική μείωση των εκπομπών και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την αλλαγή του, του κλίματος. Στην οδηγία μπορούμε να εξετάσουμε τις μέσες τιμές ανά έτος και τα διάφορα είδη εκπομπών. Δεν θα πρέπει να γίνουν κανόνας οι διάφορες εξαιρέσεις, θα πρέπει να έχουμε δείγματα κάθε έτους για να καταλήξουμε σε μέσες τιμές. Επίσης προβλέπεται η υποβολή έκθεσης κάθε δύο χρόνια, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πολύ αυστηρό μέτρο για τα κράτη-μέλη. Αν μου μένει χρόνος, θα ήθελα επίσης να εξετάσω κάποιους από τους τομείς όπου διαφωνώ με τον κύριο Γκίρεκ. αναφέρθηκε στην ανάγκη εξέτασης των χαμηλών εκπομπών. Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά. Τα κράτη-μέλη όμως θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόσουν δικά τους μέτρα για να βελτιώσουν το επίπεδο εκπομπών. Νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν μιλάμε για χαμηλές εκπομπές. Μισό λεπτό ακόμα, λέει ο Πρόεδρος. Και μία ακόμα παρατήρηση. Και έχω επίσης κάποιες παρατηρήσεις τεχνικής φύσης. Ο εισηγητής όμως ανέφερε ότι διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά για παράδειγμα τις διοξίνες και το υδρόθιο και υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί αυτές οι εκπομπές στη συγκεκριμένη πρόταση. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Έχουμε τώρα τον σκιώδη εισηγητή του ECR, τον κύριο Κροπάτσεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γκίρεκ για την έκθεσή του. Είναι μια δύσκολη έκθεση η οποία αποσκοπεί από τη μία στην ανάπτυξη και από την άλλη στην μείωση των εκπομπών. Οι εκπομπές, όπως γνωρίζουμε, αυξάνουν το κόστος. Είναι απαραίτητο όμως να εφαρμόσουμε τα μέτρα προστασίας του κλίματος ε, και να λάβουμε υπόψη την υγεία και ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το ότι η έκθεση αυτή λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία που ανέφερε ο εισηγητής. Αναφερόμαστε δηλαδή στους σημαντικούς ρήπους που έχουν συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, όπως είναι τα σωματίδια, τα, οι ενώσεις θείου, οι διοξίνες. και άλλες εκπομπές των οποίων οι συνέπειες δεν είναι απόλυτα γνωστές. Επίσης ε, τα οξύδια του αζότου είναι άλλο σημαντικό τομέα. Ε, καλύπτονται ήδη από την οδηγία για τις εκπομπές. Αφορούν όχι μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά και άλλους τομείς όπου δεν υπάρχει παρακολούθηση και έλεγχος. Η βιομηχανία πετροχημικών και επεξεργασίας ξύλου είναι σημαντικές πηγές εκπομπών. θα πρέπει η νομοθεσία να γίνει πιο σαφής, διότι έχουμε διάφορες ρυθμίσεις και διάφορες νομοθεσίες στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Συχνά δεν είναι συμβατές μεταξύ τους αυτές οι νομοθεσίες και επηρεάζουν τον ανταγωνισμό. Επίσης συχνά δεν τηρούν, τηρούνται οι νόμοι. μείωση των ρήπων στη βιομηχανία που έχουν αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία είναι απαραίτητη. Και θα πρέπει να εξετάσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να πετύχουμε μια κοινή νομική βάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ε, εκπροσωπεί την Άλντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ισηγητά για, τα... για τις προτάσεις τροπολογιών σας. Θα πρέπει να θυμηθούμε γιατί κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά. Όχι μόνο επειδή ε, έχει πλάκα να ε, εκπονούμε κανόνες για τον βιομηχανικό τομέα, αλλά για να σώσουμε ζωές. Εάν καταφέρουμε να έχουμε ένα φιλόδοξο πακέτο στο θέμα αυτό που να ευθυγραμμίζεται και με άλλες προτάσεις της Κομισιόν. Θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε από 40 έως 400 δισεκατομμύρια το χρόνο που αποτελούν τα δαπάνες για την υγεία. Και αυτό είναι μεγάλο κόστος για την κοινωνία. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό στην όλη εξίσωση. Από τη μία δηλαδή δεν θέλουμε να δυσκολέψουμε τις βιομηχανίες, από την άλλη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, το, το ποσό από τους φόρους που δίνουμε για την υγεία. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ε, τις ε, λιγότερες ε, ζημιές στην ιδιοκτησία, στο περιβάλλον, στην υγεία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ολική προσέγγιση, όχι να έχουμε υπερβολική ρύθμιση για το βιομηχανικό τομέα, αλλά να έχουμε φιλόδοξους στόχους που να ευθυγραμμίζονται με τα άλλα μέρη του πακέτου για την ποιότητα του αέρα. Θα επανέλθω με πιο συγκεκριμένες προτάσεις όταν προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να επιδιώξουμε ευρύ συμβιβασμό εντός της Επιτροπής μας, διότι όσο πιο ισχυρή είναι η θέση μας, τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε την ιδιοκτησία, των περιβάλλων και την ζωή των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία ε, ε, Ριβασί για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Καταρχάς θέλω να χαιρετήσω την πρωτοβουλία της Νέας Κομισιόν που επέμεινε από αυτό του πακέτο Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το ίδιο για τα πακέτα, για τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία. Πιστεύω ότι αυτή η οδηγία ε, θα γίνει δεκτή με πολύ ενθουσιασμό από τους πολίτες που θέλουν η Ευρώπη να προστατεύει τους πολίτες. Είναι μια οδηγία για τον ατμοσφαιρικό αέρα, αλλά στην ουσία είναι για το... την υγεία. Διότι το πρώτο αίτιο θανάτου είναι η μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα. Αυτές είναι τελευταίες πληροφορίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και από την τελευταία έκθεση του Οργανισμού Περιβάλλοντος και ε, ε, τα δύο αυτά κείμενα τονίζουν ότι στα αστικά κέντρα ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι το πρώτο αίτιο προωρών θανάτου. 80% των προωρών θανάτων και κυρίως από καρδιακά επεισόδια οφείλονται στην ε, μόλιση του ατμοσφαιρικού αέρα. Δεν είναι λοιπόν ένα μικρό θέμα. Είναι υγειονομική αναγκαιότητα να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό και αφορά φυσικά και τα οικοσυστήματα, την ε, μείωση της βιοπικιλότητας και παίζει ρόλο και στο, στην κλιματική αλλαγή θέλουμε τον ερχόμενο Δεκέμβριο να παίξουμε ρόλο στο COP στο Παρίσι. Πρέπει οπωσδήποτε να συμβάλλουμε ε, για να αντιμετωπιστεί και αυτή η πτυχή της κλιματικής αλλαγής. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολύ πιο φιλόδοξη αυτή η οδηγία, να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Όταν λέμε θα εφαρμοστεί το 2030, είναι πολύ αργά. Και οι τιμές για τους ρήπους πρέπει να είναι πολύ κατώτερες. Και να είναι πολύ κατώτερες από αυτό που τεχνικά είναι δυνατό σήμερα. Για τα ανακατομμύρια πρέπει να είναι 5, πρέπει να εφαρμοστεί ώστε να το πιο σύντομα. Γιατί αυτό προτείνει ο ΠΟΗ. Και για τις εξαιρέσεις, καλό τον εισηγητή να συμπεριλάβει, όχι να εξαιρεί τη γεωργία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί η γεωργία συμβάλλει επίσης στην ε, ατμοσφαιρική ρήπανση. Και χρειάζονται δεσμευτικέ τιμέ για ρηπαντέ που δεν συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, ο υδράργυρο. Ο υδράργυρο πρέπει να αντιμετωπιστεί στοχευμένα μετά την πρόσφατη ε, προσχώρηση στη σύμβαση του Μιναματά από την Ένωση. Και πρέπει να έχουμε και τα αναγκαία νομικά όργανα που να ε, ενθαρρύνουν θετικέ εξελίξεις που να προστατεύουν το περιβάλλον. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τις αλλαγέ. Αλλιώς στην ουσία δεν βοηθάμε ε, τους πολίτες μας που είναι εν κινδύνου. Ευχαριστώ κυρία μου, λέει ο Πώς είπατε? Παρακαλώ ανοίξτε το μικρόφωνο σας ε, πρώτα απ' όλα. Α, είστε και όλες γκουε. Α, με συγχωρείτε παραλήψη μου. κυρία Έρνστ, παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εμείς ως ομάδα έχουμε παρατηρήσεις. Φυσιολογικό. Λοιπόν, ποια είναι η σημασία αυτής της οδηγίας. Μισό εκατομμύριο άτομα αποφνίσκουν πρόωρα λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. και τεράστια ποσά, μεταξύ 277 και 900 δισεκατομμυρίων. Μπορεί να δώσει πληματικό κόστος. Άρα δεν είναι μόνο θέμα ε, ρήπανσης και περιβάλλοντος, είναι και θέμα υγειονομικό. Η πρώτη παρατήρηση για τον εισηγητή. Καλή έκθεση αυτή που υποβάλλατε. Μπορεί να αποτελέσει καλή βάση για διαπραγματεύσεις, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά μέσω συζητήσεων για να προχωρήσουμε ε, περαιτέρω. Οι τροπολογίες 8 και 11, για παράδειγμα, τις υποστηρίζουμε κατηγορηματικά. Αλλά ορισμένα άλλα πρέπει να συζητήσουμε. Για παράδειγμα, το θέμα της ευελικτοποίησης. Πρέπει να υπάρχει τέτοιος ε, διακανονισμός να βρούμε μία μέση οδό. Και είναι δυσχερές το θέμα. Και αν εξετάσουμε τους στόχους, πολλοί οργανισμοί που ασχολούνται με την υγεία και άλλοι μας είπαν ότι οι στόχοι μείωσης δεν είναι και ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Μήπως λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε την οδηγία. Αυτό είναι το ερώτημα. Πρέπει να είναι πιο φιλόδοξοι οι στόχοι, πιστεύω, να το σκεφτούμε τουλάχιστον. Και αστείο μας φαίνεται που οι ενδιάμεσοι στόχοι δεν είναι πραγματικά δεσμευτικοί. Μόνο οι τελικοί στόχοι του 2030. Αυτό είναι πολύ αργά. Δεν είναι καλό. Πιστεύω λοιπόν πρέπει να κάτσουμε να δούμε τι μπορεί ακόμη να βελτιωθεί. Πολύ καλή έκθεση, μπορεί να αποτελέσει όμω τη βάση σε πολλά σημεία για περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Έρνστ, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα για το EFDD, ποιο θέλει να πάρει το λόγο. σα ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή Κέρεκα για την εξαιρετική έκθεση. Πρέπει να πω ότι και οι συνάδελφοι, και εδώ είμαι περήφανο που είμαι σε αυτή την Επιτροπή, γιατί πραγματικά και σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, βελτιώνουμε τις υποδείξεις και τις προτάσει τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο υπάρχουν κάποια αδυναμίες. Ε, υπάρχουν δύο διορθωτικά όρια. Όπως ήδη είπαν ε, οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα, ε, καταρχήν θεωρούνται ως ε, θεωρούν ότι ο άνθρωπος επικρατεί, κυριαρχεί σε σχέση με την οικονομία. Είναι αλήθεια ότι η οδηγία ορίζει μία μείωση ε, που, των ρήπων που επηρεάζουν την υγεία κατά 70%. Όμως ο στόχος ε, αυτός ε, καθορίζεται από το κατά πόσο αυτό σημαίνει και οικονομικό κόστος. Μέχρι το 2020 δεν προβλέπεται αρκετή μείωση των εκπομπών που οδηγούν σε ασθενείες και που επιβαρύνουν τα εθνικά συστήματα υγείας και την κοινωνία ολόκληρη. Ε, προσθέτω ότι υπάρχουν εκπομπές ε, από τη γεωργία και από την κτηνοτροφία και όλα αυτά τα βλέπουμε στα παραρτήματα της οδηγίας, όλα αυτά εξαρτώνται από διάφορες πρακτικές που δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε στην ουσία το πώς παράγουμε τρόφιμα να μειώσουμε τη χρήση χημικών προϊόντων και να καταργήσουμε την εντατική κτηνοτροφία αλλά και την εντατική γεωργία. Να καταναλώνουμε λιγότερο κρέας και να ε, αναπτύξουμε την ε, γονιμότητα των εδαφών μέσω της βιολογικής ε, καλλιέργειας. Θα πρέπει να μειωθούν και οι εκπομπέ του μεθανίου, ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολείται αυτή η οδηγία. Να θυμίσω ότι υπάρχει ένα περίφημο κείμενο που λέει ότι ένα, μια γελάδα ε, ρηπαίνει περισσότερο από ένα σουβ ε, αυτοκίνητο και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Θα Υπάρχουν διάφορα σημεία που μπορούν να βελτιωθούν. Ας πούμε, η μείωση του black carbon είναι μια ανάγκη αλλά εκφράζεται σχετικά αόριστα και το αφήνουμε στην καλή βούληση των κρατών μελών. Δικαιολόγητα επίσης αποκλείονται από τον υπολογισμό των ε, εκπομπών τα νησιά, ε, τα υπερπόντια εδάφη, αλλά και τα, οι θάλασσες εκτός των ε, χωρικών υδάτων. Λες και η γη χωρίζεται σε αεροστεγή, υδατοστεγή κομμάτια. Όμως θα πρέπει να, υπάρχουν, να μην υπάρχουν περιθώρια λιγμού, είναι άσκοπα και αυτά ε, ε, οδηγούν στην ε, ελάφρυνση των υποχρεώσεων που απαιτούνται από την οδηγία. Σας ευχαριστώ. And on behalf of Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Μαριάν Βένιγκ εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές. Για λόγους χρόνου, όπως κάνετε και ορισμένοι από εσείς, θα ήθελα να θυμίσω κάποια βασικά στοιχεία και το λόγο για τον οποίο προσπαθούμε να ασχοληθούμε με κάποια από τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά ε, προβλήματα υγείας. Θέλουμε να περιορίσουμε κατά 50% τον αριθμό των θανάτων που μέχρι το 2030. Είναι σημαντικός στόχος αυτός νομίζω πέρα από τα περιβαλλοντικά ωφέλη που μπορούν να απορρεύσουν από αυτή την οδηγία. Επίση, θα πρέπει να είναι σαφέ ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρήπανση. Είναι κάτι διαφορετικό από τι κλιματικέ αλλαγέ, γιατί οι ατμοσφαιρικές εκπομπέ μπορεί να έχουν διαφορετικό αντίκτυπο ανάλογα με το πού συμβαίνουν. Επίσης ε, προσφέρουμε μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη για το πώς θα πετύχουν τους στόχους αυτούς οι οικονομικοί στόχοι είναι σημαντικοί. Ήδη αναφέρθηκαν κάποια αριθμητικά στοιχεία από κάποιον από εσάς, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, αλλά έχουμε άμεσες, άμεσα και έμεσα οικονομικά ωφέλη που ευνοούν τους πάντες, καθώς και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Γύρω στις 100.000 θέσεις απασχόλησης υπολογίζεται. Δεν θα πρέπει να το υποτιμούμε αυτό. Η Κομισιόν καλωσορίζει τη γνωμοδότηση και τις επικοδομητικές προτάσεις που έγιναν. Ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτές, για που συνέταξε την έκθεση και επίσης ακούγοντάς σας εδώ θα εξετάσουμε βεβαίως όλα αυτά τα σχόλια με περισσότερες λεπτομέρειες. Θα ήθελα ωστόσο να προβώ σε κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τα συγκεκριμένα σχόλια που διατυπώθηκαν στην έκθεση. Καταρχήν, νομίζω ότι όσον αφορά την καλύτερη ε, νομοθεσία και την παρακολούθηση, ο εισηγητής έχει ένα θέμα με τον τρόπο με τον οποίο έχει οργανωθεί αυτή η οδηγία. Δηλαδή αισθανόταν ότι δεν υπήρχε σαφήνεια όσον αφορά τα παραρτήματα, όπως τα είπε. Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πρόκειται για το σώμα της οδηγίας μαζί με τα παραρτήματα που είναι τεχνικής φύσης και είναι μια πρακτική συνηθισμένη. Είναι αλήθεια ότι εντός αυτών γίνεται αναφορά και σε άλλα έγγραφα που μπορεί να προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς. Πράγμα που ορισμένες φορές μπορεί να απαιτεί κάποια παραπάνω μελέτη. Από την άλλη πλευρά είναι επίσης απόλυτα φυσιολογικό το να γίνονται παραπομπές σε τέτοια έγγραφα. Αλλά Επίσης το να μην ενσωματώνονται όλα αυτά τα έγγραφα στη συγκεκριμένη νομοθετική πράξη. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της καταμέτρησης των εκπομπών των μικροσωματιδίων, μιλήσατε για 2,5 μικρο. Ε, πολύ μικρά είναι αυτά τα σωματίδια και επίσης αναφερθήκατε σε κάποιους άλλους ρήπους. Υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση για τα PM2,5, αλλά αυτό καλύπτει και όλα τα άλλα σωματίδια που είναι μικρότερα. Και διαβουλευτήκαμε στην προπαρασκευαστική φάση με τον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα στόχους για τα εξαιρετικά μικρά σωματίδια και η σύσταση από πλευρά του είδαν ότι θα έπρεπε να εστιάσουμε τις ε, υποχρεώσεις μείωση στα PM2,5 για τα σημεία 2 και 5 άλλη ρήπη, ε, ρωματικοί υδρογονάθρακε, διοξίνε. Εδώ έχουμε για να κάνουμε με τις μαζικές εκπομπές από πλευρά των κρατών μελών που δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα υγείας ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν ξεχνάμε τους άλλους ρήπους. Όπως γνωρίζετε, έχουμε διάφορες άλλες οδηγίες που αφορούν τις συγκεκριμένες εκπομπές, την οδηγία των βιομηχανικών εκπομπών και επίσης, για παράδειγμα, τους χλωριούχους υδρο, αρωματικούς υδρογονάθρακες. Ίσως λοιπόν ε, σε αυτή την οδηγία να μην είναι το καλύτερο σημείο για να ασχοληθούμε με αυτές τις εκπομπές. Έγινε επίσης αναφορά για, το χαμηλ... για τις εκπομπές χαμηλού επίπεδου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα βέβαια, γιατί αυτές οι εκπομπές είναι τμήμα των εθνικών εκπομπών και θα είναι κομμάτι του προγράμματος ε, ε, ελέγχου εθνικού ρήπων. Δεν σημαίνει αυτό καθόλου ότι δεν τα αντιμετωπίζουμε. Όμως, καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις συγκεκριμένες χαμηλού επίπεδου εκπομπέ είναι να συμπληρώσουμε με ε, νομοθεσία που αφορά ακριβώς ε, τις χαμηλού επίπεδου ε, εκπομπές. Έχουμε, ας πούμε, τις την οδηγία Eco Design που καλύπτει πολύ μικρές ε, εγκαταστάσεις αλλά και την οδηγία περί ποιότητας του αέρα που απαιτεί σε περιπτώσεις όπου η ρήπανση ξεπερνά τους στόχους μας να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Είτε αφορούν αυτά τις μεταφορές είτε άλλους, άλλες πηγές ρήπανσης. Αυτό το αποφασίζουν τα κράτη-μέλη. Βέβαια, οι μεταφορές είναι πολύ σημαντικές. Κάποιοι ανέφεραν το πρόβλημα που έχουμε με το ντίζελ. Και... Αλλά όπως γνωρίζετε, και αυτό είναι κάτι που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή και θα σας υποβάλουμε πρόταση για ε, τα συγκεκριμένα και Άλλο σχόλιο αφορά την επέκταση των εξάπλωση μάλλον των εκπομπών ανεξάρτητα από τα σύνορα, δηλαδή αεροπλοεία και ναυσιπλοεία. Μάλιστα, μου επιτρέπετε να αναφερθώ σε αυτά τα σχόλια. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ένα στοιχείο εδώ είναι ότι έχουμε ένα διεθνέ πλαίσιο για αυτό το είδο τη εκπομπέ και τη ρύθμιση του και άρα δεν μπορούμε άμεσα να μπούμε σε αυτά τα θέματα στη δική μα οδηγία. Ε, πρέπει να περάσουμε από το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Έχω, Έχουμε εδώ αναφέρει κάποια όρια, αλλά για χάρη χρόνου δεν μπορώ να πω στι λεπτομέρειε. Για του ε, τους ατμοσφαιρικούς να πω ότι η πιο σημαντική ρήπη σε σχέση με το αεροπλοεία όσον αφορά το διοξίδιο του θείου και το μονοξίδιο του αζότου, αυτά πιο πολύ γίνονται στο έδαφος, δηλαδή από τα λεωφορεία, όχι από τα αεροπλάνα. Τώρα, για τα ανώτατα όρια 2025. Εμείς θεωρούμε πως είναι ένα σταθμός ελέγχου στο στόχο μας της τελικής μείωσης και έχουμε πει ρητά πει ότι θα πρέπει να επιτευχθούν εκτός αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τη μη επίτευξη των στόχων αυτών. Σε αυτά σταματώ και ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μας παρουσιάσατε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης για το Περιβάλλον. Και ξαναδίνω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Άνταμ Κίρεκ. Θα του παρακαλούσα να απαντήσει στις ερωτήσεις και παρατηρήσεις που έγιναν και να απαντήσει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστηκαν διάφορες παρατηρήσεις. Και βέβαια αυτή η δουλειά αποτελεί κοινή μας προσπάθεια. Δική μας δηλαδή και της Επιτροπής για το Περιβάλλον. Η Τζούλη Γκέρλινγκ από την Επιτροπή ΕΝΒΗ είναι η συγγήτρια και η δική μας έκθεση, η δική μας γνωμοδότηση είναι απλά βοηθητική δίνει κάποιες εξηγήσει περισσότερο τεχνικής φύσης, διότι εμάς μας ενδιαφέρει η πτυχή της βιομηχανίας. Αναφέρθηκαν άλλωστε και οι ρήποι από τον γεωργικό τομέα. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν κατάλαβα αυτό που υπόθηκε σχετικά με την απόσυρση αυτής της πρότασης. Επειδή ετοιμάζονται κάποιες άλλες προτάσεις και ότι αξίζει τον κόπο να περιμένουμε τους νέους 23 στόχους. Εάν όμως περιμένουμε όπως ε, άλλωστε είπε και η Κομισιόν, θα υπάρχουν και τότε ε, νέες προτάσεις που θα προετοιμάζονται και αν περιμένουμε συνέχεια τελικά ποτέ δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε κατευθυντήρες γραμμές για την μείωση αυτών των εκπομπών. Και έτσι δεν θα μπορέσουμε να μειώσουμε και το ποσοστό θνησιμότητας που συνδέεται με την ε, ρήπανση του αέρα. Είναι τεράστιο το θέμα αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο εις βάθος και να εξετάσουμε πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και γι' αυτό δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το ολοκληρώσουμε βιαστικά. Όσον αφορά το θέμα των χαμηλών εκπομπών, δεν νομίζω ότι αυτό είναι θέμα αποκλειστικά αρμοδιότητας των κρατών μελών. Είναι διασυνοριακό το θέμα, γι' αυτό είναι και μεγάλη σημασία για την Ευρώπη. Συνδέεται το θέμα με την σωστή χρήση των καυσίμων. Έτσι λοιπόν επανερχόμαστε στο βιομηχανικό τομέα και στις ε, διάφορες ε, νέες μεθόδους κάψης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους επένδυσαν τις προσπάθειές μου. Θα ήθελα να σας καλέσω να συνεργαστούμε με την Επιτροπή ΕΝΒΗ πάνω σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 29η Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Όπως είπε ο εισηγητής, αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Ένβη. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ολοκληρώσουμε τη γνωμοδότησή μας το αργότερο τον Φεβρουάριο, διότι θέλουμε να ληφθούν υπόψη οι θέσεις μας στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κατόπιν το σημείο 8 στην ημερήσια διάταξή μας. Αντίκτυπο τη TTIP στι Ευρωπαϊκές αγορέ ενέργεια και τις Μεταποιητικές Βιομηχανίες. Παρουσίαση από τον Κουν Ράντεμάκερ. Καλό τον κύριο Κουν Ράτεμάκερς να έρθει να καθίσει εδώ και να παρουσιάσει τη μελέτη του. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου να πω ότι η Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας ζήτησε την εκπόνηση αυτής της μελέτης και το βασικό ερώτημα της Επιτροπής μας είναι πώς θα επηρεάσει η TTIP τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας και τον βιομηχανικό τομέα. Και η μελέτη προσπαθεί να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το ερώτημα. Περιλαμβάνει ανάλυση του θέματος πώς μπορεί η TTIP να βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια, για παράδειγμα, αυξάνοντας ε, την ρευστότητα στην αγορά φυσικού αερίου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και ευρύ το θέμα της συμφωνίας TTIP. Και εμείς θα επικεντρωθούμε στο θέμα της ενέργειας, των εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κύριε Μάκερ, σας καλώ να παρουσιάσετε την μελέτη σας. Είναι δυνατόν ε, να το καταφέρετε αυτό σε 10 λεπτά. Θα προσπαθήσουμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. 10 λεπτά είπατε, μάλιστα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε, όπως είπε ο Πρόεδρος, ότι είναι πολύ ευρύ το θέμα αυτό. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ασχοληθούμε με τα πιο σημαντικά θέματα. Υπάρχει... Υπάρχουν αντίγραφα της παρουσίασής μας εδώ. Φασιζόμαστε στην έρευνα που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Οι διαπραγματεύσεις ε, γίνονται κρυπτό Άρα δεν έχουμε τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων. Βαζόμαστε λοιπόν σε όλη την έρευνα που έχει γίνει αυτό. Κάναμε πολλές συνεντεύξεις και έχουμε συνεργαστεί και με πολλούς ειδήμονες για την ενέργεια και το κατασκευαστικό κλάδο. Και έτσι συντάξαμε ένα έγγραφο το οποίο δημοσίευσε λοιπόν πρόσφατα η Επιτροπή σας. Λοιπόν, θα σας κάνω μια παρουσίαση για το θέμα αυτό, τι επιπτώσεις ε, μπορεί να έχει στον ε, τομέα της ενέργειας, στο κατασκευαστικό τομέα και μετά θα έχουμε πορίσματα και συστάσεις οποίες καταλήξαμε μετά από εσωτερικές συζητήσεις. Αν εξετάσουμε λοιπόν εδώ αυτή τη διαφάνεια, διαπιστώνεται ότι το εμπορικό συζύγιο στον τομέα της ενέργειας ε, είναι θετικό υπέρ της Ένωσης. Δηλαδή, αν δούμε τα προϊόντα που εισάγονται στην Ένωση, είναι λιγότερα από αυτά που εξάγουμε. Και το ίδιο και για τις υπηρεσίες. Βλέπετε εδώ. Για προϊόντα 282-196, το ίδιο και για τις υπηρεσίες και για τις επενδύσεις. Και για τα τρία τμήματα λοιπόν του τομέα έχουμε θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Πολύ σημαντικό αυτό. Οι διαπραγματεύσεις TTIP έχουν ξεκινήσει το 2013. Ξέρετε ότι ο προηγούμενος επίτροπος ε, που ήταν αρμόδιος ε, ήθελε να καταλήξουν πέρυσι. Δεν ε, κατέστη δυνατόν, έχουν γίνει 7 γύροι διαπραγματεύσεων που ασχολούνται με διαφορετικά θέματα. Συνολικά έχουμε 23 τομείς. Και οι τομείς ε, διαπραγμάτευσης είναι πρόσβαση στην αγορά, υπηρεσίες και επενδύσεις, θέματα αριθμιστικά και άλλο ένα. Η Επιτροπή μας ζήτησε να εξετάσουμε δύο τομείς συγκεκριμένα. Πρώτον, ενέργεια, δεύτερον, κατασκευαστικό τομέας. Ε, συγγνώμη, ε, μεταπητική βιομηχανία. Αν δούμε λοιπόν τι γίνεται, θα δούμε ότι το πιο σημαντικό ενεργειακό προϊόν ε, για το εμπόριο μεταξύ αυτών των δύο εταίρων, το πιο σημαντικό προϊόν είναι ο άνθρακας. Η Ένωση εισάγει 103 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Εδώ είναι τα στοιχεία από το 2013. Και δεν εξάγουμε σχεδόν τίποτα. Οι εισαγωγές ε, άνθρακα από τις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί τα τελευταία διετία πάρα πολύ. 18% των εισαγωγών άνθρακα της Ένωσης είναι από, την Ευρω... από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε επίσης και ότι ορισμένα επεξεργασμένα προϊόντα πετρελαίου επίσης εισάγονται πολύ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τα άλλα, οι περισσότερες εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων μας από την Ένωση είναι σχετικά περιορισμένων διαστάσεων. Για τα ενεργειακά προϊόντα λοιπόν εδώ κυρίως είναι τα κατεργασμένα προϊόντα πετρελαίου και ο άνθρακας. Τώρα, δασμοί και μη δασμολογική φραγμή. Επειδή υπάρχει απαγόρευση εξαγωγής αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπάρχουν ε, δασμοί χαμηλοί μόνο κατεργασμένα προϊόντα, δηλαδή βενζίνη και δίζελ. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι ανταλλαγές, αλλά υπάρχουν και μη δασμολογικά. Είναι η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Και αυτή η οδηγία αποτελεί περιορισμό του εμπορίου ή μπορεί να αποτελέσει φραγμό στο μέλλον. Και πρέπει να συζητήσουμε αυτή την οδηγία σε σχέση με το TTIP. Για τον άνθρακα είναι μηδέν η δασμή. Τι μη φραγμό θα μπορούσε να υπάρξει και ορισμένοι αντίον του. Η κλιματική πολιτική της Ένωσης είναι πιο ανεπτυγμένη από τις ΗΠΑ όπου βέβαια ποικίλει από πολιτεία σε πολιτεία. Για τις ανανεώσιμες είναι κυρίως ε, προϊόντα αιωλικής ενέργειας και επίσης και φωτοβολταϊκά. Και οι πιο σημαντική δασμή είναι 2,7 και 1,25%. Συνολικά λοιπόν η δασμοί είναι πολύ χαμηλή. Άρα δεν θα αλλάξει πολλά το TTIP. Αλλά υπάρχουν ε, αξιόλογοι μη δασμολογικοί φραγμοί. Εκεί το TTIP θα μπορούσε να βοηθήσει. Επιπτώσεις ε, στην αγορά ενέργειας. Άνθρακας δεν έχουμε δασμούς. Οπότε όλα είναι καλά. Ακόμη και αν δεν υπάρξει TTIP, θεωρούμε ότι οι απαγορεύσει εξαγών μπορεί να επηρεαστούν από το TTIP, αλλά δεν θεωρούμε ότι θα γίνουν μεγάλες αλλαγές. Το Μεξικό και ο Καναδάς είναι μόνε εξαιρέσει για τις ΗΠΑ. Και σε όλε τις συζητήσει που γίνονται στις ΗΠΑ ε, δεν βλέπουμε να έχουν αλλάξει άποψη. Δεν υπάρχουν τάσεις ε, κατάργηση αυτών των ε, απαγορεύσεων όσον αφορά τις αγωγές από τις ΗΠΑ. Βέβαια η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων δεν επηρεάζει άμεσα. Θεωρούμε ότι θα αυξηθεί το εμπόριο σε LNG. Και, αν, ε, και αυτό θα συμβεί ιδίω εάν μειωθούν οι τιμές του φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή είναι πιο επικερδές για τις ΗΠΑ να εξαγάγουν προς την Ασία και όχι προς εμάς επίπτωση στην ενεργειακή ασφάλεια. Βλέπετε ότι λέμε πολλά εάν. Εάν καταργηθούν οι απαγορεύσει. Εάν γίνει ελκυστικό το εμπόριο. Εάν ε, συμφωνηθεί ένας μηχανισμός για αντιμετώπιση κρίσεων, τότε θα μπορούσε το TTIP να έχει θετική επίπτωση. Αλλιώς δεν θεωρούμε ότι θα έχει το TTIP ε, επιπτώσεις για την ενεργειακή ασφάλεια. Και το τελευταίο μου slide. εάν αφαιρεθεί, αφαιρεθούν οι προϋποθέσεις για, το, ε, τοπικό, για τοπική ποσόστοση, τότε θα μπορούσαν να υπάρξουν επιπτώσεις. Και βεβαίως θα μπορούσε να βελτιωθεί και ο οίκο σχεδιασμός. Είναι πιο αυστηρή νομοθεσία μας στην Ευρώπη αλλά έχει αναπτυχθεί αρκετά και ο οίκος σχεδιασμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Στέφαν Σλίεμπαντ. Είμαι συνάδελφος του Κουν Ράντεμάκερς, είμαι ερευνητής στην ίδια ομάδα και θα ασχοληθώ με τον μεταποιητικό τομέα. με αυτό είναι παρόμοια κατάσταση με τον ενεργειακό. Η δασμοί είναι πολύ λιγότερο πρόβλημα από ότι η μη δασμολογική φραγμή. Έχουμε παρουσιάσει ορισμένους τομείς, για τους περισσότερους τομείς είναι μηδέν οι δασμοί. Σε δύο τομείς όμως υπάρχουν φραγμοί είναι τα μεταποιημένα τρόφιμα και τα αυτοκίνητα. Εδώ βλέπετε όμως ότι οι μη δασμολογικοί φραγμοί έχουν ε, σημαντική διάσταση. Και σε ορισμένους κλάδους ε, είναι πολύ σημαντική αυτή η φραγμή. Συνολικά λοιπόν για τον κλάδο τι μπορούμε να πούμε ότι 80% των αναμενόμενων ωφελών από το TTIP θα προκύψουν από την κατάργηση των μη δασμολογικών φράγμων. Και συνολικά τι επίπτωση θα έχει στο μεταπητικό κλάδο. Εξετάσαμε μερικές ποσοτικές μακροοικονομικές μελέτες και το αποτέλεσμα εξαρτάται από το ποια εναλλακτική και από ποιό είναι ο συντάκτη της έκθεση, Αλλά όλα τα σενάρια δείχνουν περιορισμένη θετική επίπτωση στο ΑΕΠ τη Ένωση έω 1% αναφέρονται σε μία βασική μελέτη και μία άλλη εκτεταμένη μελέτη το εκτιμά έως και 4%. Και πού διαφέρουν οι μελέτες για διάφορα θέματα αλλά ιδιαίτερα στο βαθμό που θεωρούν το TTIP θα έχει θετικά παράπλευρα αποτελέσματα σε άλλες χώρες πέρα από τις εμπλεκόμενες χώρες. Ορισμένοι θεωρούν ότι αυτές οι παράπλευρες ε, επιπτώσεις θα είναι σημαντικές ενώ άλλοι θεωρούν ότι θα είναι μάλλον αρνητικές. Τώρα, επιμέρους τομείς. ιδιαίτερα ο τομέας ε, των μετάλλων και των ε, ηλεκτρικών μηχανημάτων και μηχανών όπου θα υπάρξουν ε, προβλήματα. Ενώ σε άλλους τομείς βλέπουμε θετική επίπτωση. Όπου θα υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επίπτωσεις δύο πρώτους. Και τι επιπτώσεις θα έχει στις διάφορες χώρες. Αντίθετα από αυτά που αναφέρονται ορισμένες φορές, ότι δηλαδή η Γερμανία θα ωφεληθεί κυρίως από το TTIP, ανάλογα, συγγνώμη, με βάση τις μελέτες, κυρίως χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Φιλανδία, Σουηδία θα αποφεληθούν κυρίως και ουσιοδός. Πού οφείλεται αυτό, Αυτές οι χώρες έχουν ε, τον υψηλότερο βαθμό εμπορίου με, την, ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και βεβαίως θα ωφεληθούν και οι χώρες που έχουν τους περισσότερους φραγμούς. Οι πολύ ήδη ανοιχτέ οικονομίες όπως οι χώρες Μπενελούξ θα ωφεληθούν σχετικά λίγο. Τώρα επίπτωση στην αγορά εργασίας. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που θα περιληφθούν στο TTIP και είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα σε τι βαθμό η μικρότερη προστασία των εργαζομένων στις ΗΠΑ θα επηρεάσει την ε, ανταγωνιστικότητα των ε, ευρωπαϊκών εταιριών διότι στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες έχουμε χαμηλότερο κόστος ενέργειας και εργασίας, ενώ στην Ένωση έχουμε περισσότερη καινοτομία, ενεργειακή απόδοση και δεξιότητες. Αλλά συνολικά θεωρούμε ότι θα είναι μειωμένες οι επιπτώσεις ε, στην ε, αγορά εργασίας. Θεωρούμε ότι μπορεί να προκύψει μισό της εκατό αύξηση απασχόλησης. Και για την καινοτομία τώρα, τελική διαφάνεια, οι εταιρείε που έχουν υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης θα ωφεληθούν περισσότερο από πρόσβαση σε ευρύτερες αγορές για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα επίμαχο είναι οι ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ περισσότερη προστασία περιφερειών από ό,τι οι Ηνωμένε Πολιτείες. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Ένα άλλο σημείο που είναι ανοιχτό, οι επιπτώσεις του TTIP στους μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης, ιδιαίτερα στο πρασίνισμα της βιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Από ό,τι κατάλαβα, ε, θα είναι στη διάθεση των μελών η έκθεση και τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η κυρία Τόια από πλευρά των Σοσιαλιστών θέλει να πάρει τον λόγο. Ναι, θέλει. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, απλά είχα σηκώσει την ε, μελέτη για να δείξω ότι την είχαμε. Δεν είναι η παρέμβασή μου προγραμματισμένη, αλλά θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να ρωτήσω το εξή. Ε, καταρχήν, Ποιος έκανε την ανάλυση για το αντίκτυπο στη μεταπητική βιομηχανία. Γιατί εκεί είναι, θα ήθελα να καταλάβω κάπως καλύτερα. Γιατί είναι αλήθεια πως λένε ότι σε περαίες περιπτώσεις όσον αφορά τον μεταπητικό τομέα δεν υπάρχουν ε, δεσμολογικές φραγμοί. Ωστόσο, όλο το έμεσο κόστος που προκύπτει από τους μη δασμολογικούς φραγμούς που είναι το ίδιο επικίνδυνοι. Θα ήθελα λοιπόν να έχω κάποια περισσότερα στοιχεία και να μας διευκολύνεται να, καταλάβουμε, να καταλάβουμε γιατί βλέπετε συχνά ακούμε ότι αυτή η συμφωνία θα άνοιγε μεγάλες αγορές και θα σήμαινε μεγάλα κέρδη για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να καταλάβω πώς θα γίνει αυτό το υπέροχο μέλλον της ευημερία και του πλούτου Μιλάτε για 5% του ΑΕΠΑ ως αύξηση, αλλά και απόλυτη για κάποιους τομείς όπως αυτός του χάλιβα, ας πούμε, της χαλιβουργίας γενικώ. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν θα ήταν δυνατόν να καταλάβουμε, αν τις απαντήσεις τις έχετε εδώ θα τις, δώσω, θα ε, κοιτάξω. Μήπως μπορείτε να μας κάνετε μια πιο εις ανάλυση για τις πτυχές του αντίκτυπου στον μεταπητικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος εξ ονόματος του ECR, μάλιστα, ο κύριος Γκοβέρντο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια σύντομη ερώτηση για την χημική βιομηχανία. Διότι το πρόβλημα είναι η ε, χαμηλή τιμή του φυσικού αερίου και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές διαφυγές από την ευρωπαϊκή παραγωγή της ε, χημικής βιομηχανίας προς την Αμερική. Διότι εκεί το, η τιμή του φυσικού αερίου είναι πολύ χαμηλότερη, ιδιαίτερα για την παραγωγή λιπασμάτων ή πλαστικών. Εσείς ε, τι πιστεύετε, τι επιρροή θα έχει το TTIP θα μπορέσει να εμποδίσει αυτή τη διαδικασία ή θα τη σταματήσει ή κάτι άλλο θα γίνει. Um, Madame Mlinar. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μίλνερ. Σα ευχαριστώ για αυτή την ε, περιστατωμένη μελέτη. Δεν έχω δει όλες τις λεπτομέρειες βέβαια ακόμα, δεν τι έχω μελετήσει. Έχω μια ερώτηση όμω. Είδα μόλι ότι είχατε μια σελίδα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω Οι μεγάλες εταιρείε δεν χρειάζονται τη TTIP. Αν πραγματικά θέλουμε να το επιδιώξουμε αυτό και εγώ πιστεύω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία, θα πρέπει να αποδείξουμε πως ε, περιέχει πλανεκτήματα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Μπορείτε εσεί να μα δώσετε μια εικόνα για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στι μικρομεσαίε επιχειρήσει αυτή η συμφωνία. κύριος Ραϊμόν, εξ ονόματος των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Είπατε ότι 103 ε, εκατομμύρια τόνοι εξάγονται ετησίως από τις ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει πιθανότητα η μελλοντική περιβαλλοντική πολιτική θα επηρεαστεί και πώς ε, σύμφωνα με την ε, TTIP. Τι σχετικές ρήτρες περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να επανέλθω στους μη δασμολογικούς ε, φραγμούς. Να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί. Είμαι νέο μέλος της Επιτροπής θα με ενδιαφέρεται να μας πείτε συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτό. Είπατε πολύ σύντομα θετικό αρνητικό. Είπατε ότι για τη μεταλλουργία και την ε, ηλεκτρική βιομηχανία υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτή η κλάδη είναι σημαντική για την περιοχή μου. Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα. Και μετά γίνεται ολόκληρη ε, συζήτηση για τη σύνδεση TTIP και κλιματικής αλλαγής. Γιατί ορισμένοι προτίθενται να εισαγάγουν σχιστολιθικό, ε, συγγνώμη, φυσικό αέριο ε, σχιστολιθικής από σχιστολιθικές άμμους. Όμως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ε, δεν ανταποκρίνεται στους ε, στόχους μας για την κλιματική αλλαγή και για τις πολύ μικρές μικρομεσαίες. Αυτές που απασχολούν μέχρι 20-30 εργαζόμενους είναι 80% των όλων επιχειρήσεών μας. Θα ήθελα να μας πείτε πώς θα επηρεαστούν. Τι θα τις ωφελήσει αυτή η συμφωνία στην πράξη. Ο κύριος Ταμπουράνο, EFDD. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον, ε, τους, τους ε, εισηγητές μας ε, και καλωσορίζουμε αυτή την έκθεση για το TTIP που μάλλον ελπίζουμε πως θα αρθεί αυτό το πέπλο μυστικότητας γύρω από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, πραγματικά θα ήθελα να έχουμε συγκεκριμένα ε, και καταμετρήσιμα αποτελέσματα. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν τους συγκεκριτές μας αν είναι βέβαιοι για τα συμπεράσματά τους. Πρώτον, εάν η αντίσταση των Ηνωμένων Πολιτειών στο να δεχτούν τις γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης που είναι η ιδιαιτερότητα του τομέα των τροφίμων της Ένωσης θα μπορούσε αυτό να επηρεάσει τη δική μας παραγωγή τροφίμων. Δηλαδή η TTIP μπορεί να θεωρήσει απλά τρόφιμα που περιέχουν γάλα, γιαούρτι και, και αλάτι σαν να ήταν απλά τρόφιμα δηλαδή όλα αυτά τα ένα σωρό τα ιταλικά και τα γαλλικά που εμείς θεωρούμε εξαιρετικά έπειτα ε, πολλές βιομηχανίες μετακινούν ε, την έρευνα και ανάπτυξη στην ΕΠΑ από την Ευρώπη, γιατί το κλίμα εκεί είναι γενικώ πιο θετικό. Τρίτο σημείο αφορά την ενέργεια. Η έκθεση λέει σαφώ ότι η TTIP δεν θα συμβάλλει στην βιομηχανοποίηση της ε, Ευρώπης, γιατί πάντα θα κοστίζει η παραγωγή λιγότερο στις ΕΠΑ. Άρα λοιπόν η TTIP δεν θα σημαίνει κανένα πλεονέκτημα όσον αφορά την ενέργεια τον εφοδιασμό ούτε για την παραγωγή πετρελαίου φυσικού αερίου, ακόμα και αν αυτή αυξηθεί στη ΣΥΠΑ. Ε, Εσεί συμφωνείτε με αυτό το συμπέρασμα. Σα ευχαριστώ πολύ. Let me also put a question before the... Before you... Να σας υποβάλω και εγώ μια ερώτηση πριν ε, να απαντήσετε γιατί πρόκειται για τον πρώτο γύρο ερωτήσεων εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων και αφορά την ενέργεια. Μισό λεπτό. Θα έχετε και δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Εγώ είμαι στον πρώτο γύρο και κάνω την ερώτησή μου εξονόματος του ΕΛΚ, γιατί είμαι εισηγητή για το θέμα. Ναι, λυπούμε, Κριστιανής, ναι, δεν το διευκρίνησα. Στο δεύτερο γύρο θα μπορέσετε όλοι να θέσετε ερωτήσεις. Μια πολύ απλή ερώτηση γιατί πρόκειται για το εμπόριο ενεργειακών αγαθών και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ισοζύγιο εμπορικό οι Αμερικανοί στέλνουν άνθρακα. Και μάλλον και εμείς θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς τον Αμερικανικό άνθρακα. Ενώ δεν συμφωνούμε για την εξαγωγή του φυσιολογικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα ήταν πολύ σημαντικό για την ασφάλεια ανεφοδιασμού που συζητούσαμε προηγουμένως. Πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα εάν δεν λυθεί με το TTIP, γιατί κανονικά θα πρέπει να λυθεί πολύ γρήγορα. Όπως υπόθηκε και για τη χημική βιομηχανία, κάνει μεγάλη διαφορά στο κόστος ε, παραγωγής. Υπάρχει μάλλον μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο κόστος παραγωγής της ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη. Μπορείτε να απαντήσετε και μετά θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Έχουμε δέκα συναδέλφους που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Να απαντήσω στην ερώτησή σας ε, και την ερώτηση για το σχιστικό, σχιστολιθικό αέριο και την χημική βιομηχανία και γενικά την ε, βιομηχανία ενέργειας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μιλάμε για σχιστολιθικό αέριο έχουμε, μια, έχουμε εκπονήσει μια ξεχωριστή μελέτη καθώς και για τη σχέση ανάμεσα στην εξαγωγή σχιστολιθικού αερίου από τις ΗΠΑ και τις δυνατότητες που υπάρχουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι, υπάρχει χαμηλότερο κόστος για τις βιομηχανίες που καταναλώνουν πολλή ενέργεια σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε δει τα τελευταία 5 με 10 χρόνια ε, την μεταφορά από ε, ε, τον άνθρακα στο αέριο στις Ηνωμένε Πολιτείε. Έχουμε λοιπόν εδώ ανταγωνισμό μεταξύ των βιομηχανιών, βιομηχανίες πλαστικών κλπ. Αυτό θα αλλάξει με την συμφωνία TTIP, μάλλον όχι. Όπως είπα και όπως εξηγείται πολύ καθαρά στην έκθεση, Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις που θα πρέπει να αλλάξουν προτού να δούμε να υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής σχιστολιθικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς θα πρέπει να λήξει, να καταργηθεί η απαγόρευση της εξαγωγής. Δεύτερον, θα πρέπει να μειωθεί η ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρίτον, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέταρτον, θα πρέπει και η αγορά να είναι ευνοϊκή. Δηλαδή, ακόμα και αν δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις, οι προμηθευτές αερίου θα κοιτάξουν να δούνε σε διεθνές επίπεδο ποια είναι η καλύτερη αγορά προς την οποία μπορώ να εξάγω το αέριο. Για το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι εύκολο με δεξαμενόπλια να μεταφερθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη ή στην Ασία. Αλλά μέσα στα τρία με πέντε επόμενα χρόνια δεν, βλέπω να, δεν προβλέπω να υπάρξουν αλλαγές. Πιο ενδιαφέρον θα ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξάγουν το αέριο προς την Ασία αντί για την Ευρώπη. Δεν βλέπω λοιπόν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές ή περισσότερες εξαγωγές αερίου από τις ΗΠΑ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφής αυτή η απάντηση. Η απάντησή μου νομίζω είναι αντικειμενική. Αν συνομιλήσετε με ανθρώπους από τον τομέα φυσικού αερίου, και εγώ από εκεί προέρχομαι, δεν νομίζω ότι θα ακούσετε άλλες απαντήσεις, διαφορετική απάντηση από αυτή που μόλις σας έδωσα. μπορούν να παρέμβουν ε, οι ευρωβουλευτές. Όχι, παρακαλώ, απαντήστε πρώτα στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ωραία, θα απαντήσω εγώ σε κάποιες από τις άλλες ερωτήσεις. Είχαμε την ερώτηση σχετικά με τους διάφορους τομείς και γι' αυτό ίσως θα ήταν χρήσιμο να επανέλθουμε στην σχετική διαφάνεια Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους διάφορους τομείς, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν προσεκτικά υπόψη. Σε διάφορες μελέτες που υπάρχουν, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι οι περισσότεροι τομείς θα επωφεληθούν. Κάποιοι τομείς όπως είναι τα μέταλλα ή οι ηλεκτρικές ε, μηχανές, τα ηλεκτρικά μηχανήματα, μπορεί να μην επωφεληθούν. Αυτό λοιπόν ίσως είναι κάτι που θα πρέπει να λάβει υπόψη της η Επιτροπή σας. Να εξετάσετε δηλαδή την ανταγωνιστική θέση αυτών των τομέων σε σύγκριση με τις Ηνωμένε Πολιτείες για να δείτε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την κατάσταση. Όσον αφορά την ερώτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μελέτες που εξετάσαμε δείχνουν ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα υποφεληθούν από τη συμφωνία TTIP. Θα έχουν στη διάθεσή τους μεγαλύτερη αγορά. Και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την έρευνα και καινοτομία. Φαίνεται ότι αυτές θα υποφεληθούν περισσότερο. τέθηκε μια ερώτηση σχετικά με τους φραγμούς, τους μη δασμολογικούς φραγμούς που υπάρχουν. Έχουμε το ευρύ φάσμα από απαγόρευση εξαγωγών μέχρι διαφορές στα πρότυπα. Πρόκειται για μια μεγάλη κατηγορία μέσων που περιγράφεται και στην έκθεσή μας. όσον αφορά την ε, γεωγραφική προέλευση. Πράγματι, διακυβεύονται οι γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω είναι δύσκολο να βρεθεί λύση σε αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλέ τέτοιε ε, γεωγραφικές ενδείξει προέλευση. οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν. Αυτό λοιπόν θα είναι δύσκολο θέμα, πιστεύω, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Όσον αφορά το χάλιβα, πρόκειται για τομέα που καταναλώνει πολλή ενέργεια. Έτσι λοιπόν επηρεάζεται από τα όσα συμβαίνουν στον τομέα της ενέργειας, όπως εξήγησε ο συνάδελφός μου ο κύριος Δεν πιστεύουμε όμως ότι θα δούμε σημαντικές εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη που αναφέρονται πότε-πότε στο πλαίσιο της TTIP. Υπάρχουν σαφώς ελκυστικότερες αγορές στην Ασία. Οι αυξημένε εξαγωγέ λοιπόν πιθανότατα να έχουν προορισμό την Ασία. Ο κύριος Ράντεμακερς, να προσθέσω κάτι σχετικά με τις ε, σχετικά με τις βιομηχανίες ε, που καταναλώνουν ε, πολλή ενέργεια. Υπάρχουν εδώ πολλές βιομηχανίες, υπάρχει βιομηχανία μετάλλων, του, του χαλκού, του ψευδάργυρου κλπ. Κυρίως έχουμε εδώ προέλευση την Ασία και άλλες χώρες και όχι τις Ηνωμένε Πολιτείε. Από εκεί προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος του ανταγωνισμού τα τελευταία δέκα χρόνια. Όταν κάνει λοιπόν κανείς προσωμιώσεις για να εξετάσει τις συνέπειες της TTIP, βλέπουμε αρνητικές επιπτώσεις για κάποιους τομείς υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν αυξημένη δυνατότητα εισαγωγής χάλιβα από τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, και ε, αυξημένης παραγωγής με χαμηλό κόστος αλλά οι δυνατότητες αυτές είναι αρκετά περιορισμένες. Αν εξετάσει κανείς τη θέση των τομέων αυτών τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ευρώπη, ε, ανταγωνιστές μας εδώ είναι κυρίως ε, η Μέση Ανατολή, η Ασία και η Ισλανδία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε μακρύ κατάλογο, ερωτήσεων, ε, μακρύ κατάλογο ομιλητών. Παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι συγκεκριμένο. Είπατε, ορισμένοι τομείς θα ωφεληθούν, ορισμένοι θα φυγούν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική αντίθεση μπορεί να είναι αν φυγεί κάποιος τομέας, χρειαζόμαστε περισσότερους φραγμούς. Η άλλη δυνατότητα, και γι' αυτό θέτω το ερώτημα έτσι, είναι σε ποιους τομείς θα ωφεληθεί η Ευρώπη και τι ποσοστού του ΑΕΠ είναι σήμερα. Ίσως αυτή είναι η τομής θα έπρεπε να είναι στο κέντρο της προσοχής μας. Είναι οι πιο παραγωγικοί τομείς της οικονομίας μας. Οι τομείς που προσθέτουν την υψηλότερη αξία, με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι είναι πολιτική η ε, επιχειρηματολογία μου. Ευχαριστώ κύριος Παολντή. Όπως ήδη είπατε, η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η TTIP δεν θα αυξήσει την ενεργειακή επάρκεια γιατί οι πόροι, οι υπά εξαρτώνται από διαφορετικά πράγματα από αυτό που περιλαμβάνει η TTIP. Δεν θα έπρεπε να αυξηθούν υποτίθεται ή ούτε οι εισαγωγές. Όμως ε, αυξάνεται η ουτε οι εισαγωγε ομως αυξανεται η ζητηση για φυσικό αέριο στις ε, στην περιοχή των χωρών Ασίας ε, Ειρηνικού. Οι στόχοι είναι πιο ενδιαφέροντες για τις κοινωνίες, τις επιχειρήσεις ε, τις αμερικανικές. Ε, εσείς είπατε ότι η αγορά είναι όρημη για αυτή την κατάσταση. Όμως, ε, ορισμένες επιχειρήσεις ήδη διαπραγματεύονται την προμήθεια φυσικού αερίου από τους προμηθευτές των ΗΠΑ. Από πού προέρχονται αυτές οι συμβάσεις οι οποίες είναι υπό εξέλιξη. Μιλάμε για μίνιμουμ κομμάτια, τμήματα ή μπορεί να είναι σημαντικά ποσοστά. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Έλερα. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι μεθοδολογική. Έχουμε ανοίξει τα μισά κεφάλαια. Και σε μεγάλο βαθμό δεν έχουμε καταλήξει σε αποτελέσματα. Με τι μέθοδο καταλήξατε ότι θα έχει έμεση επίπτωση στην αγορά εργασίας θα ήθελα να μου πείτε ποια ήταν η συλλογιστική σας. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Και δεύτερη ερώτηση. Επί του περιεχομένου. Ο συμβατικός τρόπος ε, θεώρησης των δασμών και των μη θεσμολογικών φραγμών είναι ότι Μέσω κατάργησης ε, των εμποδίων αυτών θέλουμε να υπάρξει περισσότερη ενοποίηση στην αγορά. Και θέλουμε να αναρμονίσουμε και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Παράδειγμα, τηλεπικοινωνίες. Έχουμε τα τελευταία πρότυπα στις τηλεπικοινωνίες. Εδώ και 10 χρόνια τα έχουμε συμφωνήσει. Και η Samsung θέλει να δει ποιος θα προχωρήσει ε, ταχύτερα ε, για να δει πώς θα αναπτύξει τα προϊόντα της γιατί ενδιαφέρεται για να έχει πρόσβαση ώστε να τον ε, ταχύτερα στη μεγαλύτερη αγορά θα προσαρμοστεί στα αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι ή οι Κινέζοι διότι Το θέμα που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως ε, η προοπτική, διότι τα άλλα θέματα είναι κυρίως θέμα συμβατικής ε, αντιμετώπισης των, δασμών, των φραγμών στο εμπόριο. Ο κύριος Μόιζα. Παρακολουθώ ε, ως μέλος της Επιτροπής ΙΝΤΑ στενά τα θέματα TTIP και δεν παρακολουθώ πολύ καλά, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά αυτά τα οποία είπατε για τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Βεβαίως για να εισαχθεί φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βεβαίως ε, υπάρχει αυτή η απαγόρευση εξαγωγών φυσικού αερίου, αλλά εάν υπάρχει συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, τότε αυτόματα έρονται αυτοί οι περιορισμοί. Πολλές χώρες της Ασίας δεν έχουν συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με τις ΗΠΑ. Άρα δεν είναι πλανητική η αγορά για, τη φυσική τους, ε, για το φυσικό τους αέριο γιατί έχουν και την ε, νομοθεσία τους για την ενεργειακή ασφάλεια. Το TTIP βέβαια είναι μια μεγάλη δυνατότητα εξαγωγής φυσικού αερίου και για ανταγωνισμό με την Ευρώπη. Αν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στην τιμή όπως έχουμε στις τιμές φυσικού αερίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ένωσης τότε φυσιολογικά θα έχουν κάθε κίνητρο οι Αμερικανοί να μας πουλήσουν και εμείς θα είχαμε κάθε κίνητρο να αγοράσουμε. Γιατί λοιπόν αυτό. Δεν θα συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια το θέμα των υποδομών, είναι ουσιώδες. Πρέπει να προσαρμοστούν οι σταθμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μπορέσουν να εξαγάγουν το αέριό τους. Αλλά τα υπόλοιπα επιχειρηματά σας δεν τα καταλαβαίνω. Σαβίνη. Σας ευχαριστώ. Ένα από τα πιο επίμαχα θέματα για, σε αυτή τη συμφωνία είναι το ACDS ε, καταρχήν χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση που αφορά τον αντίκτυπο της θετήψης στην ενέργεια και όχι πάντα μια συζήτηση για τα γεωργικά προϊόντα που είναι πολύ σημαντικά αλλά που στο εμπορικό ισοζύγιο δεν καλύπτουν πάνω από το 8%. Συνήθως για αυτό το πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για την TTIP. Ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την φάση ευάθεσης. Για να επανέλθουμε στο SDS όπως ξέρετε αφορά τη δυνατότητα που έχει σύμφωνα με αυτή τη ρήτρα μια εταιρεία να παρέμβει κατά των κανόνων μιας χώρας, των νόμων μιας χώρας και λέγοντας ότι ε, είναι ε, ενάντι στη διεθνή νομοθεσία αλλά αυτό ε, σε, κάποιον τρίτο, σε κάποια τρίτη δικαιοδοσία. Αυτό μπορεί να είναι πολύ περίπλοκο, ιδιαίτερα στην ενέργεια, όπου οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες είναι τεράστιες. Άρα λοιπόν το πεδίο αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κόφοντ. Thank you, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη σας. Μία ερώτηση. Αναφέρατε στην παρουσίασή σας ότι για τις ανανεώσιμες αναφερθήκατε στην αιωλική ενέργεια, έχουμε το υψηλότερο συγκριτικό πλεονέκτημα εμείς ως Ευρώπη στον τομέα της αιωλικής ενέργειας. Άρα αν καταργηθούν οι μη δασμολογικοί φραγμοί, ελπίζουμε ότι θα εξαγάγουμε, θα κάνουμε πολλές εξαγωγές στον κλάδο αυτό. Αλλά μπορείτε να μας δώσετε στοιχεία ποσοτικά. Εκεί που ηγούμεθα τεχνολογικά στις ανανεώσιμες, όχι μόνο το, την αιωλική, ή και σε πιο παραδοσιακούς ενεργειακού τομεί. Πόσο θα κερδίσουμε μπορείτε να μας δώσετε ποσοτικά στοιχεία. Αλλά και άλλη μια ερώτηση. Για τα θέματα τη αγοράς εργασίας. Πολλέ μελέτες έχουν καταδείξει ότι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας λόγω του ανταγωνισμού. Έχουμε εδώ αριθμητικά στοιχεία. Κατά πόσο θα αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων αν υπάρξουν τέτοιου τύπου μελέτες. Ε, υπάρχουν μελέτες, για παράδειγμα, στη βιομηχανία πόσο θα αυξήσει το εισόδημα. Ο Στάλφος Τουρμές. Τουρμές, μάλιστα. Ευχαριστώ για τη μελέτη. Για το φυσικό αέριο, συμμερίζομαι τις απόψεις σας. Στις ΗΠΑ είναι τέσσερα. Στο στην Ευρώπη 8, στην Ασία 15. Ε, μόλις επέστρεψε από μια σύσκεψη στο Αμπου Ντάμπι, όπου συμφωνήσαμε όλοι, ότι εάν υπάρξουν δυνατότητες εξαγωγής LNG από τις ΗΠΑ, δεν είναι πολύ πιθανό ότι θα εξαγάγουν στην Ευρώπη. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι το Κατάρ, για να μειώσει τις τιμές του αλλά γενικά συμφωνώ με την ανάλυση σας. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Οι Αμερικανοί ποτέ δεν υπέγραψαν τη χάρτα για την ενέργεια. Και έχουμε ένα νέο γύρο συζητήσεων για αυτήν την ενεργειακή χάρτα που θα πρέπει να καταλήξουν επισήμως να καταλήξει αυτός ο γύρος τον επόμενο Μάιο. Όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε για το ISDS είναι λίγο παράλογη γιατί δεν έχει υπογραφεί ακόμη αυτή η χάρτα που είναι το κυριότερο μέσο προστασίας στον τομέα της ενέργειας. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Γιατί στην ουσία είναι αντιφατικές αυτές οι συζητήσεις. Θέλουν να μας πιέσουν να δεχθούν το ISDS αλλά δεν έχουν ε, υπογράψει τον ε, πιο σημαντικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Κάπου στη μελέτη λένε, λέτε ότι το TTIP θα σημάνει περισσότερο εμπόριο πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου. Ξέρετε ότι τα δηληστήριά μας ε, αντιμετωπίζουν πρόβλημα γιατί μειώνεται η ζήτηση. Αν υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες ε, εισαγωγής ε, μεταποιημένων προϊόντων πετρελαίου στην Ευρώπη θα είναι αρνητική αντίδραση στον κλάδο. Και τέλος για τον σχεδιασμό. εάν συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς θα χρειαστεί να ρίξουμε το επίπεδό μας. Αυτό είπατε. Καλά σας κατάλαβα. Είπατε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να έχουμε συνεργασία για τον καθορισμό των προδιαγραφών γιατί θα μειωθούν οι προδιαγραφές μας. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Thank you very uh, Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο. Θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις για τη μελέτη αυτή, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θίγει μια σειρά πολύ κέριων ερωτημάτων. Άκουσα και τις παρατηρήσεις ε, των Ευρωβουλευτών. Καταρχάς θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση για την ενέργεια και για τη γενική φύση μιας συμφωνίας. Πρόκειται για εμπορική συμφωνία λοιπόν και η εμπορική συμφωνία θέτει το κατάλληλο πλαίσιο. Προσπαθούμε λοιπόν με τη συμφωνία αυτή να αντιμετωπίσουμε τους περιορισμούς που υπάρχουν από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών όταν μιλάμε για το αργό πετρέλαιο, όπου έχουμε απαγόρευση, και για το φυσικό αέριο. Μας είπαν ότι δεν είναι πολύ πιθανό να αρθεί η απαγόρευση αυτή, μια γνώμη είναι αυτή, αλλά σας περιγράφω τον στόχο των διαπραγματευτών. Βασικός στόχος λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμφωνία αυτή είναι να αρθεί η απαγόρευση εξαγωγής αργού πετρελαίου. Και όσον αφορά το φυσικό αέριο δεν υπάρχει απαγόρευση εξαγωγής. Υπάρχει όμως ε, ένα σύστημα πιστοποίησης για τους εισαγωγείς και θέλουμε το σύστημα αυτό μη αυτόματης έκδοσης πιστοποιητικών να γίνει αυτόματο όσον αφορά τις εξαγωγές προς τις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους διαπραγματεύσεις αυτές. Κάποιοι ομιλητές ανέφεραν ότι αν συναυθεί αυτή η ε, συμφωνία, τότε θα, γίνουν, ε, τότε θα γίνει αυτόματη η έκδοση των πιστοποιητικών. Αλλά παρόλα αυτά πρόκειται για προσαρμογή σε ένα σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών το οποίο δεν θα μας προστατεύσει στο μέλλον. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε λοιπόν είναι να συμπεριληφθεί μια ρήτρα στη συμφωνία που να προβλέπει αυτές τις ρυθμίσεις για εξαγωγές προς την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τι θα γίνει στην αγορά είναι ξεχωριστό θέμα από τη σύναψη της συμφωνίας. Ε, θέλουμε με τη συμφωνία να θέσουμε το πλαίσιο ώστε να διευκολυθούν οι εξαγωγές προς την Ευρώπη σε περίπτωση που αλλάξουν οι συνθήκες στην αγορά. Και νομίζω ότι υπάρχει μια σειρά ενδείξεων που δείχνουν ότι μέσω πρόθεσμα μπορεί κάλλιστα να αλλάξουν οι προϋποθέσεις της αγοράς και να γίνουν πιο ελκυστικές οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι είναι σήμερα. Βέβαια όλα αυτά εξαρτώνται και από το τι θα συμβεί στην Ασία και όσον αφορά τη θέση σημαντικών εταίρων όπως είναι η Ιαπωνία στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Θα έχουμε επανεκκίνηση δηλαδή, του πυρηνικού προγράμματος της Ιαπωνίας εξαρτάται από την ολοκλήρωση κάποιων έργων υποδομών στην Ασία που μπορεί να καταστήσουν λιγότερο ελκυστικέ τι εξαγωγέ των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ασία. Αλλά βέβαια δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι εάν η συμφωνία καταφέρει να βελτιώσει τις προϋποθέσεις εξαγωγών ε, από τις Ηνωμένε Πολιτείες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυτό θα είναι θετικό. Κάτι που δεν τονίζεται αρκετά κατά τη γνώμη μας στην έκθεση σχετίζεται με τον δεύτερο μας στόχο στις ενεργειακές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ που είναι να δημιουργηθεί ένας πίνακας κανόνων ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο που να ευνοεί τον ανταγωνισμό όσον αφορά τα ενεργειακά προϊόντα. Και αυτό το πλαίσιο δεν αναφέρεται στις δυσκολίες που έχουμε διμερώς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σχετίζεται με δυσκολίες που έχουμε με τρίτες χώρες. Όπως γνωρίζετε δεν, υπάρχουν, ε, δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς οι διεθνείς κανόνες στο θέμα αυτό. Γι' αυτό θέλουμε να δράξουμε την ευκαιρία των διαπραγματεύσεων TTIP για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Διακόπτει ο Πρόεδρος τον ομιλητή. Πρόεδρε, θα κλείσω Ευχαριστώ. Θα επισκεφθούμε την Επιτροπή σας όταν θα συζητήσετε τη σχετική γνωμοδότηση και θα σχολιάσουμε περαιτέρω. Προς το παρόν, όπως γνωρίζετε, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και προβλέπεται ο 8 γύρος κατά την εβδομάδα της Δευτέρας Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων και σε συνδυασμό με την Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ε, υποσχόμαστε ότι θα έχετε μόνιμη πρόσκληση προς την Επιτροπή μας. Παρακαλώ να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Πολύ σύντομα. Όσον αφορά τη μεθοδολογία. Στον κύριο Έλεν να απαντήσω. Είπα στην αρχή ότι δεδομένων των ε, λίγων μηνών που είχαμε για να εκπονήσουμε αυτή τη μελέτη δεν ε, έχουμε κάνει πρωταρχικές έρευνες. Δηλαδή τα νούμερα προέρχονται κυρίως από υπάρχοντα στοιχεία και από το Κέντρο ε, Ερευνών Οικονομικής Πολιτικής όπου γίνεται μια μελέτη για τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Δεν έχουμε τα αποτελέσματα των ε, διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται, γι' αυτό ε, έχουμε προσφύγει σε τέτοιες πηγές όσον αφορά τα αριθμητικά μας στοιχεία. Δεν έχουμε δηλαδή ποσοτικοποιήσει εμείς στοιχεία. Δεν ήταν δυνατόν αυτό, δεδομένου του χρονοδιαγράμματος για την φώνηση αυτής της μελέτης. Όσον αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό. Είναι σαφές ότι δεν περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαμηλώσει τα πρότυπα στον τομέα αυτών. Ακούσαμε την ερώτηση του κυρίου Τούρμες, νομίζω. Οι δοκιμές και η συμμόρφωση είναι τεράστιο θέμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμόρφωση δηλαδή με τις απαιτήσεις του οικολογικού σχεδιασμού. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών της Ευρώπης. Και πέρα από αυτό είναι σαφές ότι αν θέλουμε να εναρμονίσουμε τους κανόνες θα πρέπει να εξετάσουμε τα αποτελέσματα των δοκιμών. Οι δύο γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής που ασχολούνται με τον οικολογικό σχεδιασμό δεν έχουν σκοπό να ε, μειώσουν τα πρότυπα. Είχαμε μια συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οικολογικό σχεδιασμό, όπου στόχο είχαν να εξετάσουν ποιο θα είναι ο δρόμος στο μέλλον. Δεν έχουμε πάντως σκοπό να αλλάξουμε τα πρότυπα. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, είναι σαφές ότι τίθεται το θέμα σε τι βαθμό η κλιματική αλλαγή μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην συμφωνία TTIP. Από τη Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα και από τις άλλες γενικές διευθύνσεις που ασχολούνται με το σύστημα εμπορίας εκπομπών και άλλα, δεν είναι στόχος να αλλάξει αυτό στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας. Θα παραμείνει δηλαδή τρόπον την εμπόδιο αυτό. Αν κοιτάξετε την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, θα διαπιστώσετε ότι με τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας αυτής υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορεί να εξάγει κανείς ε, πετρέλαιο ή παράγωγα προϊόντα. Έχουμε λοιπόν ε, τρόπο να ε, ένα ε, τέτοιο εμπόδιο το οποίο υπάρχει στη συμφωνία TTIP. Και όσον αφορά το, το φυσικό αέριο, επειδή είναι ο τομέα μου θα μπορούσα να σας μιλήσω πολύ ώρα για το θέμα αυτό. Προτείνω να το κάνουμε διμερός όμως. 1,2 PCM ε, προβλέπεται για εξαγωγές ε, για τα ε, μέλη FTA, ενώ για τους άλλους προβλέπεται να είναι 1 PCM. Είναι πιο εύκολη η κατάσταση λοιπόν. Εάν έχουμε ξεχωριστή συμφωνία TTIP με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό θα είναι πλεονέκτημα στο μέλλον. Και όπως ακούσαμε από τον κύριο Τούρμες, εάν κοιτάξουμε τη χοντρική αγορά φυσικού αερίου, θα διαπιστώσουμε τεράστιες διαφορές στις τιμές ανάμεσα στις διάφορες υπήρους. Και υπό τις παρούσες συνθήκες είναι πιο ενδιαφέρον να εξάγει κανείς προς την Ασία αντί για την Ευρώπη. Αλλά αν έχετε και άλλες ερωτήσεις, ευχαριστώ, θα απαντήσω δημερός. Ευχαριστώ να προσθέσω πολύ σύντομα διότι μας έμεινε μία ερώτηση από τον πρώτο γύρο. Εξετάσαμε το θέμα της έρευνας και ανάπτυξης ε, στην μελέτη μας και δεν προβλέπεται σημαντική διαφυγή εγκεφάλων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της συμφωνίας TTIP από ό,τι, από δείχνουν οι υπάρχουσες μελέτες. Όσον αφορά τα στοιχεία για την απασχόληση, αναφερόμαστε σε αυτά πιο αναλυτικά στην ε, μελέτη μας. αλλά οι διάφορες μελέτες δείχνουν αύξηση της απασχόλησης κατά 0,5%. Αλλά βέβαια όλα αυτά εξαρτώνται από τον τρόπο υπολογισμού. Πάντως οι συνέπειες για την αγορά εργασίας ε, δεν προβλέπεται να είναι δραματικές. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και να κλείσω. Τέθηκαν κάποιες άλλες ερωτήσεις για το ISTS, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις αυτές ε, απαντώνται στην μελέτη. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις για μας, πολύ ευχαριστώ, θα σας απαντήσουμε μετά τη συνεδρίαση. Σας καλούμε λοιπόν, εάν έχετε ερωτήσεις για τη μελέτη αυτή, να... Εάν έχετε ερωτήσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν από την έκθεση, να μας τις στείλετε γραπτός. Ευχαριστώ. Κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Όπως βλέπετε είναι καυτό θέμα για την Επιτροπή μας. Θα χαρούμε να σας βλέπουμε συχνά στην Επιτροπή μας μαζί με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσβλέπουμε σε εντατικές συζητήσεις πάνω στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι για την έκθεσή σας. Και τώρα να περάσουμε στο σημείο 9. Μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δάση και για τους ε, τομείς ε, δασοκομείας. Μια νέα λοιπόν στρατηγική για τα δάση για τον δασικό τομέα. Πρόκειται για γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Γεωργίας που είναι η αρμόδια επί επιτροπή. Ο εισηγητής μας είναι ο Μάρκ Ιώζεφ Γκρουμπάζικ. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο για να μας παρουσιάσετε τη γνωμοδότησή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ η γνωμοδότηση που έχουμε στέξει αφορά, αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δάση και το τομέα της υλοτομίας και της δασοκομείας. Τα δάση είναι πολύτιμος ε, κοινωνικός ε, και οικονομικός ε, τομέας. Πολλές φορές μάλιστα αποτελούν τμήμα της εθνικής κληρονομιάς που ελέγχεται και συντηρείται από το κάθε κράτος. Πρόκειται για ένα κληροδότημα και για τις επόμενες γενναίες. Για αυτούς τους λόγους θα πρέπει να φροντίζουμε πολύ ε, το συγκεκριμένο τομέα. Όσον αφορά τον οικονομική πτυχή, τα δάση αποτελούν το 40% της επιφάνειας της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επιφάνεια αυτή αυξάνεται κατά 0,44% ετησίως βέβαια από όσον αφορά γενικότερα τον υπόλοιπο κόσμο, οι δασικές εκτάσεις μειώνονται. Επίσης, ε, στα δάση απασχολούνται 3,5 εκατομμύρια κόσμος. σημαντικό μεγέθη δηλαδή όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή δεν είναι ε, σκληρή νομοθεσία πρόθεση έχει να δημιουργήσει ένα δίκτυο επαφών και να χρησιμοποιήσει τις καλύτερες δυνατές πρακτικές στη διαχείριση των δασών. Η γνωμοδότησή μας περιλαμβάνει κάποια σημαντικά στοιχεία. Καταρχήν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και την παροχή κινήτρων για την ε, ανάπτυξη στο πλαίσιο αυτής της κρίσης και της ευρωπαϊκή Πολιτικής για την Οικονομική Ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Είναι επίσης σημαντικό ζήτημα ε, από περιφερειακή άποψης, διότι σε περιφέρειες που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν, σε κάποιες μάλλον περιφέρειες δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η μηχανία, ενώ η δασοκομεία ναι και είναι πολύ σημαντική για τις τοπικές κοινότητες, όπως ας πούμε στο πλαίσιο θέσεων απασχόλησης για τους νέους, ο τομέας της δασοκομείας τους, δείχνει, ε, τους δίνει τη δυνατότητα να απασχοληθούν και να αναπτυχθούν. Επίσης, πρόκειται για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων, του κατάλληλου περιβάλλοντος, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε όσο γίνεται περισσότερα από την δασική οικονομία, καθώς και να ε, αντιμετωπίσουμε διάφορα κλιματικά ζητήματα. Θα πρέπει να θυμόμαστε επίσης τη κλιματική πολιτική, στην οποία τα δάση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και στην απορρόφηση διοξιδίου του άνθρακα ε, και θα έπρεπε να είναι ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα. Ωστόσο θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορισμένη επιρροή στην ε, δασική πολιτική καθώς αυτή εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορές καθώς και τις διαφορετικές προτεραιότητες των διαφόρων κρατών μελών. Ωστόσο, εάν το δούμε το θέμα αυτό Συνολικά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, οργανωτικά αλλά και χρηματοδοτικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις απειλές στα δάση. Φωτιές, παράνομη υλοτομία και αρρώστιες των ε, δέντρων, των δασών. Κυρίες και κύριοι, οποιοδήποτε σχόλιο είναι πρόσδεκτο και σας ευχαριστώ για τις τροπολογίες που μου έχετε ήδη στείλει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά για την έκθεσή σας. Ε, έχουμε να ακούσουμε τους κοιόδης εισηγητές. Παρακαλώ όχι πάνω από δύο λεπτά γιατί ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κυρία Βυρκόνα, εξονόμαστε το του ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Κρόμπατσεκ για την πολύ καλή γνωμοδότηση που συνέταξε και για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για αυτή τη στρατηγική είναι ότι η δασοκομεία είναι μάλλον η δασοκομεία από οικονομικής άποψης και πώς αυτός ο τομέας μπορεί να επηρεάσει θετικά την απασχόληση. Δεν πρόκειται μόνο δηλαδή για προστασία των δασών, ε, η πολιτική δασών είναι κάτι το οποίο εμπίπτει ε, στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, θα πρέπει να παραμείνει και εδώ έχουμε ένα πλεονεκτικό στοιχείο γιατί πρέπει να τονίσουμε το ρόλο των δασών στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών μπορούμε να επωφεληθούμε από τα δάση με βιώσιμο τρόπο ε, ως δεξαμενές άνθρακα να τα χρησιμοποιήσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δάση και τη βιομάζα των δασών ώστε να προωθήσουμε την αυτάρκεια στην ενέργεια. Θέλαμε να υπάρξει περιορισμός της γραφειοκρατίας, αυτός είναι πολύ σημαντικός στόχος γιατί δεν αφορά μόνο την ανταγωνιστικότητα αλλά και την παραγωγή νέων προϊόντων, υπηρεσιών, αλλά και την προώθηση και την κατασκευή σπιτιών με ξύλα στην Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό εδώ. Για να γίνουν όμως όλα αυτά δυνατά, θα πρέπει να εστιάσουμε στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Που είναι ένα σημαντικό τμήμα το οποίο δεν αναφέρεται εδώ. Όσον αφορά την ψηφιακή Ευρώπη, θα θέλαμε να έχουμε κοινή Ευρώπη εδώ στο νοσοκομικό τομέα διότι υπάρχει κοινή βάση δεδομένων για τη νοσοκομεία και είναι πολύ σημαντικό. Η κυρία Κουμπούλα Νάτρη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Γκρουμπάτσικ για την πολύ καλή ε, γνωμοδότηση της, ε, που ετοιμάσατε για την Ήτρε. Και επειδή η Ήτρε είναι ε, βιομηχανία έρευνα και ενέργεια, έχουμε άμεση σχέση με τα δάση και θα πρέπει να αναλάβουμε την πρόκληση της, χαμηλής, της οικονομίας χαμηλού άνθρακα στην Ευρώπη ή να δούμε και την βιοοικονομική πτυχή της στρατηγικής για τα δάση. Επίση, όλα αυτά συνδέονται με την ανάγκη για δημιουργία θέση απασχόληση και εξάλλου ο τομέα τη δασοκομεία αυτή τη στιγμή παρέχει δουλειά σε 3 εκατομμύρια Ευρωπαίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίση υπάρχει και όλη η αλυσίδα των αξιών. Τώρα, η δικευμένα εργατικά χέρια είναι βασικά για την δασοκομεία όπως και για τη βιομηχανία και καλά εκπαιδευμένο εργατικά, εργατικό δυναμικό χρειάζεται. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να πείσει ε, τους ανθρώπους να, πείσουν, ε, να δουλέψουν στην εξοχή ε, γιατί οι πόλεις προσελκύουν τους νέους. Γι' αυτό και γίνονται, μάλλον αν γίνουν προτάσεις τέτοιου τύπου από κοινού ε, στην Ευρώπη, θα βοηθήσουν στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Δεξαμενή άνθρακα και απορρόφηση διοξιδίου του άνθρακα μπορούν να αποτελέσουν τα δάση, αλλά μπορούν να μειώσουν και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, τις ε, δύο εκπομπές και πρέπει όλα αυτά να τονιστούν και από την Επιτροπή Έρευνας υπάρχει ψηλή προστιθέμενη αξία και ε, δυναμικό ανάπτυξης ε, για χρήση ξυλίας στις οικοδομές αλλά και στην κατασκευή δρόμων. Υποστηρίζω λοιπόν την ιδέα αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης που θα λέει ότι οι αρμοδιότητες και τα συγκεκριμένα μέτρα για αυτό το τομέα εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Εσενίκ. Ευχαριστώ. Έλεγα ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο αντιμετωπίζει τα άτομα ως μακροοικονομικές μεταβλητές. Αυτό κάνει και με τα δάση. Τα δάση δεν είναι μόνο πηγή για ξυλία και βιομάζα είναι ε, οικότοποι για τα ζώα μας, είναι οι φραγμή κατά της κλιματικής αλλαγής και παίζουν ε, ρόλο κλειδί σε βιολογικούς κύκλους όπως του ύδατος και του άνθρακα που είναι αναγκαία. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να σκέφτεται πώς θα υπερασπιστούμε αυτή μας την κληρονομιά και όχι μόνο την εμπορική εκμετάλλευση. Για να το κάνει αυτό πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο περιβαλλοντικής ε, προστασίας και να τεθεί τέρμα στην επιταχυνόμενη ιδιωτικοποίηση γιατί φαίνεται ότι 60% των δασών μας είναι ήδη σε ιδιωτικά χέρια και στην Πορτογαλία για παράδειγμα είναι πάνω από 90%. Σήμερα λοιπόν πρέπει να τονίσουμε ότι είμαστε η μέγιστη εισαγωγή του αποτελέσματος της ε, αποψήλωσης ε, των δασών του κόσμου. Και αυτό αποτελεί ε, παράγοντα τεράστιας αύξησης της παραγωγής διοξιδίου του άνθρακος. Πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι έχουμε ευθύνε και για αυτά που συμβαίνουν στα δάση και πέραν των συνόρων μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για τους πρασίνους. Όχι. Η e FTD. Α, ο κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ. Το σχέδιο έκθεσης. Πολύ καλό, ισορροπημένο. Και βεβαίως ε, είναι ενθαρρυντικό το ότι κάθε έτος αυξάνονται κατά μισό της εκατό τα ευρωπαϊκά δάση. Φαίνεται ότι τα αξιοποιούμε με καλό τρόπο. Και αυτό είναι καλό και για το περιβάλλον και για την κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα να ηρεμήσουν αυτοί που λένε ότι πρέπει να ασχολούμεθα όλο και περισσότερο με τα δάση. Βεβαίως κάνουμε πολλές προσπάθειες να συμπεριληφθούν στο εμπόριο διοξιδίου του άνθρακα. Γίνονται προσπάθειες από ορισμένα κράτη-μέλη να υιοθετήσουμε αυτή την προσέγγιση. Αλλά ας κάνουμε μια, ένα παραλληλισμό με την ε, γεωργική πολιτική. Τι θα σήμαινε να έχει αρμοδιότητα για τα δάση ένωση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κοινή εκμετάλλευση των δασών. Αν συμπεριλάβουμε τα δάση στο ε, εμπόριο στο εμπόριο της, ε, του διοξείδου του, του άνθρακα αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα, πώ θα πρέπει να γίνει ένα δάσο τι είδη δασών, τι είδη δέντρων θα φυτευτούν κτλ. Δηλαδή θα γραφειοκρατικοποιηθεί η, η ευρωπαϊκή πολιτική, η πολιτική μας για τα δάση όπω η γεωρική πολιτική. Βεβαίω όλα αυτά που λέτε για ανταλλαγή ε, εμπειριών και πρακτικών κτλ. Αλλά παρακαλώ όχι νέα νομοθετήματα, όχι νέες νομοθετικές αρμοδιότητες ε, για τα δάση της Ένωσης. Πρόεδρος. Ο Σνάφος Φρίντριχ. Με συγχωρείτε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Αυτό ήμουν σε άλλη επιτροπή. Και πρέπει να δούμε συγκεκριμένα τι αρμοδιότητες έχει η Ένωση. Πρέπει να δηλώσουμε σαφώς ως Κοινοβούλιο για το πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση των δασών. Είναι θέμα των κρατών μελών και όχι της Ένωσης. Αλλά Για παράδειγμα η έρευνα για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δάση, πώς πρέπει να διαχειριστούμε τα δάση. Γιατί δεν το ξέρουμε. Για παράδειγμα μπορούμε να κάνουμε σεντόνια από τα δάση που τα πουλάει το IKEA. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και ιδιαίτερα στην Ήπεθρο. Επίσης πρέπει να μειωθεί η άσκοπη γραφειοκρατία πολλά δάση είναι μικροεπιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να τις ε, φορτώνουμε με γραφοκρατία. Επίσης υπάρχουν ε, δυνατότητες πράσινης ανάπτυξης να παραγάγουμε περισσότερα από τα δάσημα, δάση μας. Στη Σουηδία και τη Φινλανδία τώρα έχουμε περισσότερα δάση από ό,τι είχαμε πριν από 3-4 δεκαετίες. Και παρόλα αυτά παράγονται περισσότερα από τα δάση τώρα και μειώνουμε και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ε, προωθούμε και την τηλεθέρμανση. Και έχουμε και δυνατότητες με αυτόν τον τρόπο μέσω χημικών βιομηχανιών να αντικαταστήσουμε τα ορυκτά καύσιμα με πιο βιολογικά καύσιμα. Θα υποβάλω πιο συγκεκριμένες προτάσεις για να τονίσουμε περισσότερο την έρευνα, να βρούμε νέες δυνατότητες να σεβαστούμε την επικουρικότητα και κάτι τελευταίο που πρέπει να συμπεριληφθεί δεν θα αποφασίσουμε εμείς τι θα κάνουν οι διοκτήτες δασών με τα δάση τους. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς σε ποιον θα πρέπει να πουλήσει αν θέλει ένας ιδιοκτήτης δασών το δάσος του. Ωραία. Τώρα ο εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Ιγνάθιο Σεωάνε από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργία. Τμήμα ματάρχης. Ο Ιγνάσιο Σεωάνε δεν μπόρεσε να έρθει. Είμαι ο Τόμας Έλακα από την μονάδα του. Ευχαριστούμε για την ε, θαυμάσια εργασία σας, τα σχόλια. Θα δούμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Και προσβλέπουμε στην τελική εκδοχή του κειμένου σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ο πρόεδρος. Οπότε, κύριε Σιγητά, ήδη σας επένεσαν τόσο πολύ που μπορώ να σας δώσω το λόγο. Φυσικά καλό να υπέρξει περαιτέρω συνεργασία, λέει ο εισηγητής, για να Φυσικά λοιπόν ελπίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Κύριε Σιγητά. Και τώρα η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 29 Ιανουαρίου 12 το μεσημέρι. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε στη συζήτηση και να σας ενημερώσω ότι σε μερικά λεπτά θα αρχίσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Αύριο, ως συνήθως 9 η ώρα και αύριο το απόγευμα στις 3. Έχουμε τέσσερις συντονιστές των, τέσσερα, των τεσσάρων μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων. Αλλά δεν είναι εδώ η πράσινη, η γκουε και το EFDD. Περιμένουμε λοιπόν λίγα λεπτά. Και όλοι όσοι δεν προβλέπετε να συμμετάσχουν στην συνεδρίες των συντονιστών, παρακαλώ να αποχωρήσετε ησύχως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Θα τα πούμε αύριο για άλλες 7 ώρες συνεδρίας.